So, wir freuen uns natürlich, dass Wim van der Kamp wieder gesund ist und bei uns ist. που ο Βίμ Βαντεκάμπ ανέρωσε. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε. Σας καλωσορίζω στην ε, συνεδρίασή μας. Αν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Ωραία, κανείς δεν έχει αντίρρηση. Έγκριση των πρακτικών αν δεν υπάρχει και εδώ πέρα καμία αντίρρηση, τις 15 και 16 Φεβρουαρίου επίσης εγκρίνονται. Ωραία. Περνάμε λοιπόν στο πρώτο σημείο. Παρουσίαση του κανονισμού της ΕΑΖΑ, της πρότασης ε, της Κομισιόν για έναν ε, κανονισμό για την υπηρεσία της ε, ασφάλειας αεροπορίας. Όπως θυμάστε το Δεκέμβριο η Κομισιόν είχε κάνει την πρότασή της. Εν τω μεταξύ υπάρχει και εισηγητής ε, για να περάσουμε στις ε, λεπτομέρειες του πακέτου. Λοιπόν, θα δώσω πρώτα απ' όλα τον λόγο στον κύριο Κορνέλιους από τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών για 10 λεπτά και μετά στον συνάδελφό μου τον κύριο Μαρινέσκου. Όχι, όχι τώρα, όχι τώρα, ο κύριος Κορνέλιος πρώτος από την Κομισιόν. Έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ πέρα για να σας παρουσιάσω τους ε, νέους, την πρόταση μας για νέους κανόνες για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας για τους οποίους είμαστε υπερήφανοι. Έχουμε ήδη διαφάνειες, να περάσουμε στη δεύτερη. Λοιπόν, γιατί πρώτα απ' όλα κάνουμε αυτή την πρόταση. Θεωρούμε πως είναι αναγκαίο και χρήσιμο να επικαιροποιήσουμε την υφιστάμενη νομοθεσία που υπάρχει εδώ και 10-15 χρόνια για να προετοιμάσουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο της ασφάλειας αεροπορίας για τις προκλήσεις των επόμενων 10-15 ετών. Για να είμαστε έτσι σε θέση για να συνεχίσουμε να έχουμε ασφαλείς ε, αερομεταφορές και φιλικές προς το περιβάλλον για τους ε, επιβάτες ε, και για το γενικότερο κοινό. Λοιπόν, η πρότασή μας ταιριάζει με τις προτεραιότητες της Κομισιόν και το πρόγραμμά μας για ανάπτυξη και δουλειές. Επίσης για την εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς να γίνει πιο οδηγή για την ενίσχυση της βιομηχανικής μας βάσης στον αεροδιαστημικό τομέα και βεβαίως μια από αεροπορία είναι μια ένας κλάδος παγκόσμιο, σκοπεύουμε να ενισχύσουμε και τον παγκόσμιο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αρχές που εφαρμόσαμε κατά την αναθεώρηση είναι οι εξής. Πρώτα απ' όλα, δεν θέλαμε να υπάρξει μια επανάσταση, αλλά μια εξέλιξη σταδιακή, δηλαδή να εδραιώσουμε όλα τα θετικά που είχαμε τόσα χρόνια στο υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο, παραδείγματο χάρη η λειτουργία της ΕΑΖΑ για να αναφέρω μια πτυχή. Δεύτερον, η αρχή άλλη που ακολουθήσαμε είναι ότι προσπαθήσαμε ο κανονισμός να γίνει πιο αναλογικός, να απλοποιηθεί όπου αυτό είναι δυνατόν, με το να εστιάσουμε παραδείγματο χάρη στους πραγματικούς κινδύνους και να καταλήξουμε σε μια προσέγγιση η οποία θα προσανατολίζεται περισσότερο στα αποτελέσματα και όχι στις διαδικασίες. Ένα άλλο σημείο της αναθεώρησης είναι ότι θέλαμε να ενισχύσουμε την φιλοσοφία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού συστήματος που θα εμπλέκει όλους τους ε, φορείς σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο κρατών μελών. Επίσης να δούμε την αλληλεπίδραση μεταξύ διαφόρων πολιτικών, ασφάλεια και περιβάλλον, ασφάλεια από κακόβουλες ενέργειες και από ατυχήματα. Προσπαθήσαμε επίσης να έχουμε περισσότερη ευελιξία από ό,τι στο παρελθόν για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις μελλοντικέ ε, εξελίξεις στις αγορές και στην τεχνολογία και βέβαια να έχουμε ένα κανονισμό ο οποίος θα είναι ουδέτερος ως προς την τεχνολογία και φιλικός προς την καινοτομία. Πρώτα απ' όλα, για τον στόχο του να χρησιμοποιούμε καλύτερα τους πόρους που έχουμε. Ένα από τα στοιχεία που έχουμε είναι να έχουμε μια εργαλειοθήκη για το πώς θα μπορούμε να μοιραζόμαστε τους πόρους μας ως μέρος αυτού του ενιαίου συστήματος μεταξύ των εθνικών αρχών αεροπορίας ε, μεταξύ τους αφενός και με την ΕΑΖΑ αφετέρου να χρησιμοποιούμε αυτό το οποίο λέμε τους Ευρωπαίους επιθεωρητές ε, αεροπορίας σε ένα πλαίσιο για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων έτσι ώστε η δουλειά ή η εποπτεία της ασφάλειας να λαμβάνει χώρα στον οργανισμό εκείνο και στην τοποθεσία εκείνη που είναι καταλληλότερο να γίνει. Επίσης υπάρχει ένας μηχανισμός εποπτείας ανάγκης γιατί γνωρίζουμε πως ε, το ευρωπαϊκό σύστημα κατά κάποιον τρόπο εξαρτάται από τον πιο αδύναμο κρίκο και άλλα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αναλάβουμε δράση εκεί όπου υπάρχουν κάποια κένα. Και αυτό κατά την άποψή μας ε, θα πρέπει να είναι μια ευρωπαϊκή αντίδραση στις ανεπάρκειες. Εξού και η πρόταση αυτή για ένα μηχανισμό εποπτεία ανάγκη, το οποίο φαντάζεστε βέβαια ότι είναι επίμαχο στα κράτη-μέλη. Ένα άλλο θέμα είναι ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα μήτρο πληροφοριών το οποίο θα ε, περιέχει πληροφορίες για την πιστοποίηση και την εποπτεία. Ξέρουμε πως οι πληροφορίες είναι διασπαρμένες μεταξύ κρατών μελών και ΕΑΖΑ και δεν υπάρχει έτσι σωστή εποπτεία. Οπότε στο μέλλον σκοπεύουμε να υπάρχει ένα καλύτερο πλαίσιο για ανταλλαγή αεροιατρικών δεδομένων. Και βεβαίως τώρα που είναι και η επέτειος της συντριβής της της German Wings είναι και επίκαιρο. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν πιστοποιημένοι ιδιωτικοί φορείς. Έχουμε τώρα ένα καλύτερο και ευρύτερο πλαίσιο για την χρήση αυτών των πιστοποιημένων φορέων. Επίσης είναι πιο ξεκαθαρισή απαιτήσει ε, των αρμοδίων αρχών ε, και από την ΕΑΖΑ στον νέο κανονισμό και όσον αφορά και την πιστοποίηση και τα προσόντα των επιθεωρητών που θα πρέπει να έχουν το ίδιο υψηλό επίπεδο σε ολόκληρη την Ένωση και να μπορούν να εφαρμόζουν τις ίδιους κανόνες με τρόπο ομοιόμορφο. Επίσης προσπαθήσαμε οι κανόνες να γίνουν πιο αναλογικοί για να υπάρχει ένα διαφανές πλαίσιο για εξαιρέσεις και μέτρα εκτακτού ανάγκης. Και βεβαίως, σημαντικό επίσης, στον τομέα της αεροπορίας είναι το τι συμβαίνει στον ΙΚΑ, τον Διεθνή Οργανισμό. Προσπαθούμε λοιπόν να ακολουθούμε τις παγκόσμιους ε, κανόνες και για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί ως Ευρωπαϊκή Ένωση στον ε, ΙΚΑ έχει σαχθεί εδώ πέρα ο μηχανισμός του δικτύου των ειδικών που συνεργάζονται στα παγκόσμια φόρα και βεβαίως όπως είπαμε ένα μητρό πληροφοριών ε, ρυθμιστικών διαφορών μεταξύ ημών και του ΙΚΑΟ. Τώρα, υπό τον τίτλο ενός συστήματος ευέλικτου το οποίο θα βασίζεται στα αποτελέσματα, στην απόδοση, έχουμε ξεκάθαρες αρχές για να γίνει η εξελόγηση κινδύνου. Για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε, όπως είπα, ένα κανονισμό που θα βασίζεται στην απόδοση. Ο κανονισμός λοιπόν εστιάζει περισσότερο εκεί όπου θεωρούμε ότι υπάρχει ο σοβαρότερος κίνδυνος ή η σοβαροτερη ανάγκη για μια δημόσια παρέμβαση για την ασφάλεια δηλαδή στις ε, ε, εμπορευματικές ε, αερομεταφορές, τις πτήσεις τις εμπορικές. Έχουμε πολύ περισσότερες δυνατότητες για τις εταιρείε για να επιδείξουν ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις, π.χ. Διευρύνονται οι δυνατότητες ε, να δεχτούμε δηλώσεις συμμόρφωσης, όπως σε άλλους κλάδους. Επίσης, απλοποιήσαμε τους ορισμούς, διαφορετικές κατηγορίες λειτουργίας και αεροσκαφών έχουν απλοποιηθεί, όπως και η δυνατότητα της μίσθωσης μεταξύ εταιριών, κάτι το οποίο αποκτά και όλο και μεγαλύτερο ρόλο. Υπάρχει και, υπάρχουν και άλλες δυνατότητες ευελιξίας. Τα κράτη-μέλη μπορούν να επιλέξουν το ευρωπαϊκό σύστημα για κρατικά αεροσκάφη, στρατιωτικές δραστηριότητες ή Κατασκευαστές επίσης ε, μπορούν να επιλέξουν το σύστημα αυτό για κάποια μικρά αεροσκάφη τα οποία αυτή τη στιγμή εξαιρούνται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες αλλά μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να το θεωρήσουν χρήσιμο να έχουν πιστοποιητικό της ΕΑΖΑ. Μεταφέραμε επίσης ε, στο κείμενο αυτό τις απαιτήσει του ΙΚΑΟ για την διαχείριση ασφαλείας ε, που είναι πρόσφατη εξέλιξη στο πλαίσιο του ΙΚΑΟ. Επίσης τυποποιήθηκε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Ασφάλεια της Αεροπορίας ε, και προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε την δομή του κειμένου και να εισαγάγουμε πιο τυποποιημένη ορολογία. Κάποια ζητήματα έχουν εξελιχθεί. Βεβαίω ή παρατηρήσαμε ότι δεν ε, τα κάλυπτε επαρκώς ο υφιστάμενος κανονισμός Γι' αυτό ακριβώς εδώ πέρα ενισχύσαμε το πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την αλληλεπίδραση μεταξύ των κανόνων ασφαλείας, των κανόνων για τα αεροσκάφη αφενός και τις άλλες τεχνικές πτυχές όπως η ασφάλεια από κακόβουλες ενέργειες και οι περιβαλλοντικοί κανόνες. Η κυβερνοασφάλεια επίσης ξεκάθαρα πλέον ε, αποτελεί ρόλο της ΕΑΖΑ και θα υπάρχει καλύτερη συνεργασία με την Ομοθεσία Περιχημικών Ισιών, τον οργανισμό REACH. Ένα κενό το οποίο παρατηρήσαμε ότι υπήρχε είναι η διαχείριση των υπηρεσιών εδάφους, οπότε η ανάλυση της ασφάλειας έχει δείξει πως υπάρχουν πολλά περιστατικά με, την, με τις υπηρεσίες εδάφους, οπότε αποφασίσαμε να το καλύψουμε με τον κανονισμό βεβαίως όχι με ένα δυσκίνητο πλαίσιο αλλά με ένα αναλογικό πλαίσιο. Οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις επίσης για τα αεροναυτικά προϊόντα όσον αφορά τον θόρυβο της εκπομπές ε, υπήρχαν ήδη στον προηγούμενο κανονισμό αλλά τώρα έχουν ενσωματωθεί στην ε, διαδικασία έγκρισης ε, τύπου των αεροσκαφών και έχουμε και κάποιες ε, απαιτήσει για περιβαλλοντική πιστοποίηση. Και τέλος, ένα μεγάλο κενό το οποίο είχαμε, το οποίο δεν μπορούσε κανείς να προβλέψει πριν από 10 χρόνια, είναι τα μη επανδρομένα αεροσκάφη και έχουμε εδώ πέρα ένα άρθρο, ένα παράρτημα με κάποιες διαδικασίες για να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα ασφαλείας και κυκλοφορίας μη επανδρομένων αεροσκαφών. Προτείνουμε λοιπόν οι περιορισμοί που υπήρχαν στον κανονισμό να φύγουν, που έλεγαν πως ε, όλα τα αεροσκάφη κάτω των 150 κιλών δεν καλύπτονται από τον κανονισμό. Προτείνουμε να διαγραφεί αυτό εντελώς και να έχουμε κοινού κανόνες ε, για όλα τα μη επανδρομένα αεροσκάφη ε, και το σκεπτικό είναι πως ε, η ρύθμιση θα είναι αναλογική με τους κινδύνους. Οπότε οι κανόνες δεν θα είναι οι ίδιοι για πολύ μικρά μη επανδρομένα αεροσκάφη όπως με αυτούς που θα είναι για μεγάλα επανδρομένα αεροσκάφη που πετάνε σε μεγάλο ύψος ανάμεσα στα επιβατικά. Πρόκειται λοιπόν για μια νέα προσθήκη. Ε, αν θέλετε μπορούμε να επανέλθουμε σε αυτό με λεπτομέρειες. Επίσης προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε κάποιες πτυχές ε, της ε, διοίκησης της ε, ΕΑΖΑ. Ξέρετε πως είναι μια υπηρεσία που έχει δημιουργηθεί στον κανονισμό αυτόν. Κάποιες άλλαγες στα κείμενα αφορούν την κοινή προσέγγιση που βασίζεται στην κοινή δήλωση Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Κομισιών για το πώς οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες θα πρέπει να λειτουργούν και να διαρθρώνονται. Έχει εισαχθεί ο μηχανισμός ενός εκτελεστικού συμβουλίου. Για, τις καθημερι... για την καθημερινή λειτουργία υπάρχουν νέες μορφές εσόδων, επιδοτήσεις, επιδοτήσεις από τους προϋπολογισμούς της αναπτυξιακής βοήθειας που μπορεί να χρησιμοποιήσει η ΆΖΑ για να βοηθήσει την ασφάλεια στην Αφρική ή σε άλλα τμήματα του κόσμου και για να μπορέσει να βελτιωθεί αυτή η ασφάλεια και προτείναμε να προσθεθεί επίσης η δυνατότητα ε, για νέα τέλη που θα καταβάλλονται στην ΕΑΖΑ για τη δουλειά που κάνουν για τον κανονισμό ATM και για την εποπτεία του ATM. Φυσικά θα πρέπει ε, να βοηθήσουν κάτι μελη ε, στο Eurocontrol για αυτή τη δυνατότητα χρέωσης τελών. Και μπορώ βεβαίως να σας δώσω και περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα αυτό. Έχουμε προσθέσει και διάφορους δείκτες ή ε, εμπασπιδός υπάρχει ανάγκη να αναπτυχθούν δείκτες ε, ούτω ώστε η υπαρχει αναγκη να καθορίζει το φόρτο εργασία, την αποτελεσματικότητά τη και να είναι η βάση για πιθανή αύξηση τη ευελιξία ε, σε ό,τι αφορά τον αριθμό του προσωπικού και για το πώ χρηματοδοτούνται. Ε, το ζητάει ο κλάδο να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα να προσαρμόζεται ο αριθμό των υπαλλήλων στη ζήτηση. Και πιστεύουμε ότι με βάση αυτού του δείκτε μπορεί αυτό να γίνει στα πλαίσια της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού. Και προτείνουμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε καλύτερη χρήση της πραγματογνωμοσύνης της ΕΑΖΑ σε τομείς, τέλος πάντων να δώσουμε τη δυνατότητα η Κομισιόν να ζητάει την ΕΑΖΑ να τη βοηθάει ε, με τεχνική πραγματογνωμοσύνη σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, το περιβάλλον, την έρευνα, την κατάρτιση ή την εφαρμογή του, του ενιαίου ουρανού. Και εδώ μια διαφάνεια για τα τα αεροσκάφη, όπως σας είπα, δείχνει τη διαφορά ανάμεσα στο παρελθόν και στο μέλλον, με όλες αυτές τις νέες εφαρμογές που θα γίνουν δυνατές όταν τα drones αυτά μπορούν να πετάνε πιο ελεύθερα στον αέριο χώρο μας. Η πρότασή μας είναι όλα τα ανεπάνδρωτα σκάφη να ενταχθούν στο πλαίσιο, να έχουμε κοινούς κανόνες που θα βασίζονται στο κίνδυνο και οι κανόνε θα είναι ανάλογοι με τον κίνδυνο και ανάλογοι με τον κίνδυνο τη επιχείρηση. Όχι μόνο το μέγεθο του σκάφου, αλλά και γιατί το χρησιμοποιούμε. Γιατί ξέρετε, ανάμεσα στην, στο να χρησιμοποιούμε ένα drone ε, στο κέντρο Βρυξελών ή στην βόρεια Σουηδία, Φερρυπίν. Επίση, μια σαφή διαίρεση των καθηκόντων ε, για τα ανεπάνωτα σκάφη σε ό,τι αφορά την ΕΑΖΑ και τι εθνικέ αρχέ, και διάφορε διαδικασίες θα πρέπει να προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητε των σκαφών αυτών, γιατί εδώ μιλάμε για ένα τεράστιο στόλο και πολλοί από αυτού που χειρίζονται τα drones δεν είναι συνηθισμένοι στους κανόνες τη αεροπλοεία. Και επίσης τα κράτη-μέλη ζητούν καλύτερα εργαλεία για τον έλεγχο και την εποπτεία και την εφαρμογή. Και τα σκάφη, ας πούμε, θα πρέπει ε, στο μέλλον να μην πετάνε πάνω από περιοχές που δεν πρέπει να πετάνε και χάρη σε αυτούς τους κανόνες θα μπορέσουν τα κράτη-μέλη να βοηθηθούν και να εφαρμόσουν αυτούς τους κανόνες. Ε, να εφαρμόσουν ε, αυτά που χρειάζονται. Αυτά για τα νεπάνθρωτα σκάφη και με αυτά, Πρόεδρε, κλείνω και την παρέμβασή μου. Ευχαριστώ. έμαθα να Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την παρουσίαση. Αυτό ο κανονισμό είναι πολύ σημαντικό, είναι σαφέ. Και περιμένουμε, περιμέναμε εδώ και καιρό τον κανονισμό αυτόν. Δυστυχώ στο μεταξύ ένα κατέπεσε, αλλά βλέπω ότι αυτό ο κανονισμός είναι και ισορροπημένο και ήταν αναγκαίο για τον κλάδο. Έχω κάποιε ερωτήσει. Καταρχά γιατί η Κομισιόν παρετήθηκε από την ιδέα του, e του να ονομάσει την αρχή αυτή EAA, European Aviation uh, Authority, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Αεροπορίας. Για, για μένα επίσης στην έκθεση αυτή το μεγαλύτερο, το πιο σημαντικό θέμα είναι τα ανεπάνδρωτα αεροσκάφη. Γιατί αυτά τα αεροσκάφη θα είναι, αλλά είναι ήδη μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ευρώπη. Γιατί μπορούν να κάνουν τα πάντα. Και είναι μια τεχνολογία που δεν ελέγχουμε πια. Είναι παντού. Ακόμα και στα καταστήματα παιχνιδιών, στο κέντρο της πόλης. Θα έχουμε πολλά προβλήματα με αυτά τα αεροσκάφη. Η Άζα ασχολείται, υποτίθεται, με την ασφάλεια στην αεροπορία. Παράλληλα, εδώ έχουμε να κάνουμε υπτάμενα αντικείμενα. Επομένως, θα πρέπει να έχουμε σκληρότερους κανόνους, κανόνες και θα φύγει διατάξεις στον κανονισμό για τα ανεπάνδρωτα. Αυτό θα γίνει μέσω κατεξιοδότηση πράξεων, σωστό. Αλλά νομίζω ότι οι πιο σημαντικές αρχές θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον κανονισμό. Υπάρχουν κάποιες διατάξεις που αφορούν την καταχώρησή τους. Πρέπει να απαγορεύεται να πετάνε πάνω από ορισμένε περιοχές, αλλά θα πρέπει να είμαστε ακόμα πιο σαφείς και να δώσουμε πιο λεπτομερείς απαντήσεις ε, για το θέμα αυτό. Μία ερώτηση τώρα για τα τέλη και τις κυρώσεις. Υπάρχουν δύο νούμερα, 4% ε, και 2,5%. Πώς στάσατε σε αυτά τα νούμερα κομισιών. Γιατί αν μιλάμε για μια εταιρεία που κερδίζει, που έχει κάνει τζίρο, εν πάση 50 δις, το να πληρώνει 2,5% ας πούμε του τζίρου της, φέρει πιν η Airbus. Μα θα φτάσουμε σε πολύ ενδιαφέρουσες καταστάσεις. Ακόμα και αν κάναμε μεγάλα λάθη, για να δούμε, θα το πληρώσω το 2,5% ασφάλεια. Ποια θα είναι η επίπτωση της εμπτοκής της ε, ΕΑΖΑ στον τομέα της ασφάλειας. Ειδικά σε ό,τι αφορά την κύβερνο ασφάλεια. Τι πρόθεση έχετε εδώ. Η διεθνή συνεργασία, πολύ σημαντική. Ελπίζω η ΆΖΑ να μας εξασφαλίσει την ε, ε, αμοιβαιότητα, ειδικά μεταξύ ΆΖΑ και FAA, ειδικά για τις δραστηριότητες πιστοποίησης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τον κλάδο. Θα μειωθεί έτσι το κόστος και η γραφειοκρατία, πιστεύω. Αυτά από πλευράς μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκαμπρίλε Πόισεν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή για τη σημερινή παρουσίαση. Χαιρετώ το γεγονός πως έγκαιρα έχουμε τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις για αυτό το τόσο αποφασιστικό χαρτοφύλακα, θέτοντας έτσι αποφάσεις για το μέλλον της αεροπορίας μας και συνεπώς επίσης για το μέλλον πολλών θέσεων εργασία υψηλής κατάρτισης στην Ευρώπη. Είναι γενικά αναγνωρισμένο γεγονός πως η ΆΖΑ από την ίδρυσή της κάνει πολύ καλή εργασία στον τομέα της ασφάλειας Υπάρχουν ωστόσο πολλέ αμφιβολίες σε πολλού εκπροσώπου συμφερόντων, εάν θα πρέπει να το κάνει επίση για τον τομέα τη ασφάλεια, καθώ πρέπει να λάβουμε υπόψη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση οι απαιτήσει ασφάλειας είναι πολύ μεγάλες και θα αυξηθούν στο μέλλον. Σε αυτόν τον τομέα βλέπω ωστόσο διχογνωμία, παραδείγματο χάρη μεταξύ Επιτροπής και ΑΖΑ και αφετέρου μεταξύ πολλών αεροδρομίων και κρατών μελών σχετικά με το μέχρι πού πρέπει να φτάσουν οι αρμοδιότητες της ΕΑΖΑ. Παραδείγματο χάρη θα μπορούσε να μιλήσει, να θίξει το ζήτημα των πτήσεων πάνω από περιοχέ σύγκρουση. Εδώ ένα πιο ευρύ ρόλο τη ΕΑΣΑ μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω περισσότερων πληροφοριών από τι υπηρεσίε ασφάλεια των κρατών μελών, το οποίο δεν γίνεται επαρκώ έω τώρα. Πιστεύω πω συμφωνούμε όλοι πω σε μια διασυνοριακή περιοχή πρέπει να, να επιδιώξουμε ευρωπαϊκέ λύσει Ωστόσο πρέπει να υπάρξει ένας λογικός καταμερισμός εργασιών και όχι να διπλασιάζονται οι φυστάμενες και καλά λειτουργούσες δομές. Υπάρχουν διατυπώσεις όπως η συνεργασία χωρίς να ορίζονται σαφώς. Οπότε αναρωτιέται κανείς πού θα βρίσκονται οι αρμοδιότητες στο μέλλον. Πώς θα συμπεριφερθεί η Επιτροπή ως προς αυτό. Πέραν του τομέα τη security υπάρχουν ζητήματα πιστοποίησης. Πολλά από αυτά έχουν νόημα και πιστεύω ότι εδώ στις διαβουλεύσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να μιλήσουμε περισσότερο και να κάνουμε περισσότερο για τα κοινωνικά πρότυπα. Μπορώ να φανταστώ πως τα κοινωνικά πρότυπα και η τήρησή τους πρέπει να γίνουν μέρος της ΕΑΣΑ. Τίθεται όμως και το ερώτημα Ποιε ικανότητε, τι αρμοδιότητε θα έχει η ΆΖΑ. Θέλω να τονίσω πω λόγω τη ταχεία αλλαγή στην αεροπορία και λόγω των επερχόμενων εργασιών τη ΕΑΖΑ δεν θα πρέπει να αναλογιστούμε μειώσει του προπολογισμού, καθώ έχουμε να κάνουμε με μια σειρά δρόντων η οποία φτάνει από τα αεροδρόμια ω του κατασκευαστές. Γι' αυτό και τα σχέδια για μια ευελιξία του προπολογισμού είναι απολύτω απαραίτητα. εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει να ξεκονομήσει πόρου εκεί που δεν πρέπει, βλέποντα τον εαυτό τη. Το ερώτημα όμω είναι επαρκεί το μοντέλο αυτό και θα είναι η ΕΑΣΑ ικανή να ανταποκριθεί στα καθήκοντά τη. Ωστόσο δεν βλέπω ιδιαίτερο ενθουσιασμό σχέδια που υπάρχουν, υπάρχουν εναλλακτικέ για μια διαρκή χρηματοδότηση. Και τέλος το ερώτημα του διεθνούς ρόλου της ΕΑΣΑ. Πιστεύω πως είναι λογικό πως η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ηγετική δύναμη στον τομέα της αεροπορίας χρειάζεται μια ΕΑΣΑ η οποία μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτόν τον ρόλο σε διεθνές επίπεδο. Στον τομέα της ασφάλειας έχουμε επιτύχει πολλά στον τομέα της αεροπορίας, γι' αυτό πιστεύω πως θα πρέπει να είμαστε πιο αποφασιστικοί και να δραστηριοποιηθούμε και σε διεθνές επίπεδο, περνώντας στην εξαγωγή των προτύπων ασφάλειάς μας για να βοηθήσουμε και άλλες περιοχές στην επιταξή της ασφάλειας. Και γι' αυτό θα βοηθήσουμε την ΕΑΣΑ με τα απαραίτητα μέσα, η κονδύλια, αλλά το ζήτημα δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι η πολιτική υποστήριξη, η οποία εμπεριέχει και την βοήθεια της ΕΑΣΑ σε όλα τα διεθνή φόρουμ, έτσι ώστε να αποκτήσει ένα εύλογο κύρος. Εδώ με ενδιαφέρει η εκτίμηση της Επιτροπής πόσο προσωπικό και σε ποιες θέσεις θα χρειαστεί η ΆΣΑ για να μπορέσει να ανταποκριθεί στον ρόλο της. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πέτερ Φοντάλεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, Οπωσδήποτε θα δούμε σε βάθος αυτές τις ε, προτάσεις ε, ως, ε, ως και ο Συμφωνώ πως με τον εισηγητή. Η κατάσταση όσον αφορά τα μη επανδρομένα αεροσκάφη είναι πάρα πολύ σημαντική όσον αφορά τον κίνδυνο που μπορούν να αποτελέσουν για την αεροπορία. Είχαμε, είχα και εγώ προσωπικά ένα περιστατικό με μια προσγείωση στη Γαλλία όπου απευθύνθηκε μια σύγκρουση την τελευταία στιγμή. Ένα άλλο κλασικό ερώτημα προς την Κομισιόν είναι η σχέση μεταξύ της ΕΑΖΑ και των εθνικών υπηρεσιών εποπτείας ε, της αεροπορίας. Υπάρχουν εδώ και χρόνια, τώρα μας λέτε πως οι αρμοδιότητες τους θα πάνε στην κολονία και η θέση τους εξασθενεί συνεχώς η ποιότητα των επιθεωρητών ε, είναι πάρα πολύ καλή παρόλα αυτά. Οπότε τι θα κάνετε ακριβώς ε, για την σχέση αυτή μεταξύ ΕΑΖΑ και τις αρμοδιότητες των εθνικών επιθεωρητών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ματέσα Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήδη αναφέρθηκε το θέμα των μη επανδρομένων αεροσκαφών και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι το αντιμετωπίζουμε σε αυτή την πρόταση. Έχω όμως κάποιες ερωτήσεις προς την Κομισιόν, κάποια πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα. Στο παράρτημα 9 λέει πως θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα πρόσωπα αυτά τα οποία χειρίζονται τέτοια αεροσκάφη και να υπάρχει μια εκπαίδευση. Τι θα κάνει η Κομισιόν, σκοπεύει να φέρει μια πρόταση για ομοιόμορφη εκπαίδευση αυτών των ε, ανθρώπων. Επίση, ε, θα πρέπει, όπως είπα, να μην πληγεί εδώ πέρα η αγορά εργασία όσον αφορά την εκπαίδευση των λεγόμενων χειριστών μη επανδρομένων ε, αεροσκαφών. Το δεύτερο, το ανέφερε και η συνάδελφος, αφορά τις πτήσεις πάνω από περιοχές συγκρούσεων μας αφορά και εμάς στην Ολλανδία ειδικά μετά την καταστροφή με την ε, MR70 την πτήση πάνω από την Ουκρανία θα πρέπει λοιπόν εδώ πέρα να έχει ένα σημαντικό κεντρικό ρόλο η ΆΖΑ και να υποχρεωθούν οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών να μοιράζονται τις ε, πληροφορίες που έχουν ε, να κάνουν συστάσεις ή και να λάβουμε και κάποια μέτρα ίσως για να αποφευχθούν τέτοιες καταστροφές στο μέλλον. Γιατί λοιπόν η Κομισιόν δεν κάνει κάποια ισχυρότερη πρόταση προς αυτή την κατεύθυνση για να έχουμε δηλαδή ασφάλεια και από κακόβουλες ενέργειες. Αυτά από μένα για την ώρα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Κίλνεν. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξεκινώ από την εξής βάση. Ότι το πιο σημαντικό πάντα είναι η ασφάλεια. Από εκεί ξεκινάμε. Αυτή είναι η αφετηρία μας. Αν υπάρχει ασφάλεια, ε, όλα μπορούν να λειτουργήσουν. Έχουμε αρκετά παραδείγματα στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τις καινοτόμες λύσεις. Γι' αυτό θέλω να κάνω εξή ερώτηση στην Κομισιόν. Δεν ξέρω ότι τώρα που αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα νέα προϊόντα και τις καινοτομίε, αν είμαστε στο ύψο των περιστάσεων, ε, οι θεωρήσει, ο έλεγχος, ε, η εποπτεία είναι πραγματικά στο επίπεδο που πρέπει. Και αν σε πολιτικό επίπεδο ε, είμαστε σε θέση να παρακολουθήσουμε αρκετά αυτέ τι καινοτομίε. Αυτή είναι μια αμφιβολία που έχω. Σε ό,τι αφορά την πίεση χρόνου που έχει η ΕΑΣΑ και υπό την οποία εργάζεται, αν αυτό επηρεάζει την ικανότητά της να αναπτύξει διαδικασίες έξυπνες, τυποποίησης, να ανταποκριθεί στις ανάγκες ε, και επίσης μπορεί να δημιουργήσει πολλή προβλήματα στη διεθνή, πολλά προβλήματα στη διεθνή συνεργασία, παραδείγματος χάρη συνεργασία με τις ΗΠΑ και με τον Καναδά και τον υπόλοιπο κόσμο. Κομισιόν, πώς βλέπετε το μέλλον της ΕΑΣΑ υπ' αυτή την άποψη, δηλαδή ο κόσμος αλλάζει συνεχώς. Και οι δικοί μας οι πολιτικοί, ας πούμε, κινούνται με το ρυθμό της χελώνας. Πώς μπορούμε να επιταχύνουμε αυτή την πορεία, ούτω ώστε η ΕΑΣΑ να είναι στο ύψος των περιστάσεων και να ανταποκρίνεται σε ένα κόσμο ο οποίος αλλάζει συνέχεια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Κομισιόν, λέει κυρία Αντελή, μας έδωσε πληροφορίες και μας είπε ότι η εναέρεια κυκλοφορία θα, μέχρι το 2020 θα αυξηθεί κατά 50%. Τίθενται δύο βασικά ερωτήματα. Πρώτον, ε, σε μια τέτοια αύξηση είμαστε προσαρμοσμένοι σε ό,τι αφορά τα θέματα ασφάλειας. Θα πρέπει ο κανονισμός να δώσει σε αυτή τη νέα υπηρεσία καλά εργαλεία για να εξασφαλίσει την ασφάλεια. Και δεύτερον, στο σημερινό πλαίσιο κατά πολέμηση κλιματική κλιματικής αλλαγής μπορούμε να επιτρέψουμε μια τέτοια αύξηση κατά 50% των εκπομπών ας πούμε. Φυσικά η απάντηση είναι όχι, είναι αρνητική. Όμως ο τομέας ε, της αεροπορίας ε, εκπέμπει απίστευτα ε, αέρια του θερμοκηπίου και είναι το 3% των παγκόσμιων εκπομπών. Δηλαδή ό,τι εκπέμπει συνολικά η Γερμανία. Επίσης, το δεύτερο σημαντικό θέμα του, του κειμένου αυτού είναι το περιβάλλον. Είπατε μια φράση όταν μας περιγράφετε το οργανόγραμμα. Μας είπατε το, ότι το περιβαλλοντικό θέμα θα το προτάξουμε και ότι θα εφαρμόσουμε τα περιβαλλοντικά θέματα. Θα υπάρξει πραγματικό συντονισμός ε, στο οργανόγραμμά σας σε συντονισμό με την Eurocontrol για τα περιβαλλοντικά. Φερρυπίν. Δεύτερο ερώτημα, που για μένα είναι σημαντικό, για το, τη σημασία του περιβαλλοντικού σκέλους. Εγκύπτεται επί των κανόνων, επί των, και, ε, των ε, τεχνολογικών καινοτομιών, ε, καινοτόμων καυσίμων κτλ. Έχετε δηλαδή ε, μια μακροπρόθεσμη θεώρηση, παραδείγματος χάρη όλα τα θέματα που συνδέονται με την κατανάλωση της κυροζήνης. Μιλάτε για τέλη. Δεν μπορούμε να έχουμε εναλλακτικά σενάρια ε, τιμολόγησης της ε, Δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Κάτι άλλο που μου φαίνεται επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι η ΕΑΖΑ πρέπει να εξασφαλίσει καλύτερα τα κράτη-μέλη ε, εποπτεύουν την φυσική και ψυχολογική υγεία των πιλότων. Θα πρέπει να δείτε την έκθεση για, το ατύχημα της German Wings στις Γαλλικές Άλπεις, όπου βλέπουμε ότι τηρήθηκε σε γη ηχθείως εκεί πέρα. Υπάρχει πρόβλημα ε, σε σχέση με το θέμα αυτό. Υπάρχει αυτό το κοινωνικό θέμα βέβαια, αλλά υπάρχει και το θέμα της ε, ποιότητας του αέρα, ας πούμε, μέσα στην άτρακτο και στις καμπίνες των πιλότων, ε, που υποτίθεται ότι είναι ένα θέμα που θα πρέπει να απασχολεί στην ΕΑΖΑ. Και να τελειώσω με μια άλλη ερώτηση. Πώ θα μειώσετε τις συγκρούσει συμφερόντων στο εσωτερικό αυτή τη νέα υπηρεσία τη ΕΑΖΑ. Των νέων καθηκόντων, αν θέλετε, τη ΕΑΖΑ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ τους ε, ομιλητές για την παρουσίαση που μας έκαναν. Κυρίως ε, τον εκπρόσωπο της ΕΑΣΑ. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση που θέλω να θέσω. Το κοινωνικό θέμα που συνδέεται με την ασφάλεια. Σε ποιο βαθμό θα είναι θέμα με το οποίο θα ασχολείται η ΕΑΣΑ, ούτω ώστε ατυχήματα όπως αυτό το φρικτό ατύχημα της German Wings να αποτρέπονται. Και επίσης η έκθεση που έγινε για το ατύχημα αυτό δείχνει ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και επίσης κάτι άλλο, λέμε ας πούμε για τα νεπάνδρωτα αεροσκάφη, λέμε ότι εκεί δεν υπάρχουν άνθρωποι, αλλά ναι υπάρχει ένας άνθρωπος που τα χειρίζεται από το έδαφος ας πούμε. Άρα ο ανθρώπινος παράγοντας είναι σημαντικός. Ε, ακόμα και για τα στρατιωτικά αεροσκάφη είναι σημαντικό ανθρώπινο παράγοντα. Ε, ποιοι είναι λοιπόν, ποιο είναι ο ανθρώπινο παράγοντα, Είναι οι πιλότοι και το πλήρωμα του αεροσκάφου. Όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία συνδέονται, α πούμε, με την πίεση, με την οικονομική πίεση, με την κατάσταση, α πούμε, λόγω των ορών πτήση, με τι άδειε κτλ. Όλα αυτά τα θέματα είναι άθλια στην Ευρώπη, είναι στο επίπεδο του τρίτου κόσμου. Θα πρέπει Αντί τα βελτιώσουμε, θα πρέπει να τα βελτιώσουμε. Και εμεί αντί να τα βελτιώνουμε, τα επιδεινώνουμε. Μην ξεχνάμε λοιπόν ότι οι πιλότοι επηρεάζονται από όλα αυτά τα πράγματα. Από τι ώρε πτήση και τα λοιπά. Και άρα και η ασφάλεια επηρεάζεται. Άρα θα πρέπει να κάνουμε κάτι συγκεκριμένο. Ε, συμφωνώ επίση ε, με αυτό που είπατε για την ομάδα ε, των επιθεωρητών. Και, το θέμα, και με το θέμα της κυβερνοασφάλειας, γιατί ε, έχουμε όλο και πιο περίπλοκα αεροσκάφη, όλο και πιο περίπλοκα και ξέρετε ότι ο αδύναμος κρίκος της αλυσίδας αυτής είναι σε αυτή την, ε, τα τόσο περίπλοκα ηλεκτρονικά είναι ακριβώς το θέμα της ε, κυβερνοασφάλειας. Αυτοί οι, οι εμπειρογνώμονες που θα δικτυώνονται όπου υποτίθεται θα πρέπει να συντονίζονται για να δίνουν μια γνώμη. Τι ε, επίπτωση να έχουν σε δύο βασικά στοιχεία. Πρώτον, ε, στο να δρομολογήσουμε ε, τα νέα καύσιμα, εναλλακτικά καύσιμα, δηλαδή τα οποία προέρχονται από την κυκλική οικονομία. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, με ποιον τρόπο θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τον τρόπο ε, που διαλύονται τα αεροσκάφη και παροπλίζονται τα αεροσκάφη για να μην δημιουργούν προβλήματα στο περιβάλλον. Τέλος, η ΕΑΣΑ έχει πετύχει συμφωνία με τη γερμανική ε, κυβέρνηση για την έδρα τη. Γιατί δημιουργεί αρκετή ανησυχία αυτό το θέμα. Ε, το θέμα των εδρών δηλαδή των διαφόρων υπηρεσιών και οργανισμών. Θέλουμε μετά από τόσα χρόνια να ξεκαθαριστεί η θέση της ΕΑΣΑ στην κολονία. Ευχαριστώ πολύ. Βιν Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. θεωρώ πως με την ΕΑΖΑ και τον νέο κανονισμό έχουμε εδώ πέρα αυτό το οποίο λέμε στα Ολλανδικά φοβερές δυνατότητες ανάπτυξης, ένα διαμαντάκι και θα έλεγα πως ε, το θέμα εδώ είναι ο προπολογισμό της ΕΑΖΑ, στο και αν δεν συμφωνώ πλήρω με τον εισηγητή, γιατί αν δώσουμε πολλές ε, αρμοδιότητες στην νέα αυτή υπηρεσία και ο κύριος Κορνέλισεν, ο οποίος μας είπε τόσα πολλά πράγματα για την διοίκηση και τα τέλη και τα έσοδα, ε, καλό θα ήταν νομίζω να μας πει η Κομισιόν, Συμβούλιο και η Συγητής τι γίνεται με τον προϋπολογισμό. Αν δηλαδή το, αν το συγκρίνουμε με τον προϋπολογισμό της ε, Αμερι, Αμερικανικής FAA. Μιλάμε για Γολιάθ και Δαβίδ. Εντάξει μπορεί ο Δαβίδ να είναι πιο έξυπνος. Ε, ναι και κερδίζει το τέλος, ναι το ξέρω. Αλλά δούμε και τον ερευνητικό προπολογισμό της ΕΑΖΑ. Είναι πάρα πολύ περιορισμένος, ε, ειδικά αν έχουν καινές αρμοδιότητες. Θα ήθελα να δω πώς επηρεάζει αυτό τον προπολογισμό τους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Λούση Άντερσεν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Λίγα πράγματα να σας πω. Πρώτα απ' όλα ανησυχώ βλέποντας ε, την αξιολόγηση αντικτύπου και το σχέδιο του κανονισμού για το ότι η Κομισιόν δεν έχει δώσει ιδιαίτερο βάρος στους εργαζόμενους ε, των αεροπορικών εταιριών, πιλότους και λοιπούς, που ανησυχούν για το ότι δεν απαιτείται πλέον το ίδιο επίπεδο πιστοποίησης χωρίς ε, να παρέχονται εδώ πέρα τα απαραίτητα στοιχεία. Πρόκειται για έναν τομέα κρίσιμο για την ασφάλεια όπως γνωρίζουμε και συμφωνώ εδώ πέρα ε, με το ότι η Κομισιόν σε μεγάλο βαθμό ξαναγράφει τους ε, στόχους, ε, παραδείγματο χάρη να αυξάνονται οι απαιτήσει περιβαλλοντικής προστασίας. Αλλά η ασφάλεια πρέπει να είναι το πρώτο και κύριο και θα ήθελα να μάθω κάποια περισσότερα πράγματα. Επίσης, για το θέμα των συνθήκων εργασίας και αξιοπροπών στις εργασίας, ε, της επαρκούς εκπαίδευσης, ε, ε, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι η μεταχείριση του προσωπικού δεν θα επηρεάσει αρνητικά την ασφάλεια. Για μένα το σχέδιο αυτό απλά δεν τα λαμβάνει υπόψη επαρκώς αυτά τα ζητήματα. Σας ευχαριστώ. Μάισνερ. Ευχαριστώ. Από τις μια σύντομη ερώτηση έχω προς την Κομισιόν αφορά την ασφάλεια και συμφωνώ εδώ πέρα με τον συνάδελφο που ανησυχεί για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Εμένα απασχολεί κάτι άλλο, το λέω πάντα. Το ADSP, τα μεγάλα αεροσκάφη έχουν συστήματα αναγνώρισης αμοιβαίας και τηρούν αυτομάτως τις ε, αποστάσεις ε, και είναι πάρα πολύ θετικό αυτό αλλά είναι ακριβές συσκευέ που δεν τις έχουν τα μικρά αεροσκάφη και από όσο έχω μάθει εκπέμπουν σε διαφορετικές συχνότητες ε, για μένα αυτό μπορεί να είναι ένα πρόβλημα ασφαλείας πριν από λίγους μήνες υπήρχε μια σύγκρουση μεταξύ ενός τζάμπο και ενός μικρού ιδιωτικού αεροσκάφους στην Αφρική Θεωρώ λοιπόν πως είναι πρόβλημα και δεν υπάρχει τίποτα εδώ πέρα στον κανονισμό. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε ναι, να υπάρχει καινοτομία με συστήματα τα οποία ασφαλείας τα οποία θα αναγνωρίζει το ένα το άλλο, αλλά οτιδήποτε κινείται στον αέρα, μεγάλο ή μικρό, θα πρέπει να έχει μία συχνότητα που θα εκπέμπει για να βλέπουμε τι κινείται πού. Νομίζω πως απαιτείται κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ Γιάννης Νίλσεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. δύο ερωτήσεις. Είχα τελικά απέμεινε μία, γιατί με κάλυψαν οι συνάδελφοι. Αφορά το θέμα των συνθήκων εργασίας. Το δεύτερο μου ερώτημα λοιπόν αφορά μια γενικότερη πτυχή. Η εντολή της ΕΑΖΑ μας λέτε ότι θα ενισχυθεί ε, και υπάρχουν όλο και περισσότερα πράγματα τα οποία αναλαμβάνει η Ευρώπη και οι ευρωσκεπτικιστές μας λένε πως ε, τώρα έχουμε άλλον έναν υπερεθνικό οργανισμό που θα ασχολείται με την ασφάλεια των πτήσεων και αυτό σημαίνει πως χρειάζεται μια πολύ ισχυρή εντολή. Ας δούμε π.χ. την Σουηδία και την Εστονία. Είναι δύο κράτη-μέλη και ας υποθέσουμε ότι στην Σουηδία δίδεται μια σύμβαση σε μια αεροπορική εταιρεία και μετά υπάρχει ένα συμβάν. Και λένε οι Σουηδικές αρχές, ναι εμείς θα ελέγξουμε το αεροσκάφος και πιθανώς θα παγορεύσουμε τις πτήσεις. Αλλά δεν μπορεί η αρχή αυτή να λάβει αυτή την απόφαση γιατί είναι ένα εστονικό αεροσκάφος και δεν μπορεί να λάβει αυτή την απόφαση μόνο της Σουηδίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να πούμε πως υπάρχουν δύο αρχές που μπορεί να έχουν διαφορετικά συμπεράσματα και θα υπάρχει κάποιος, ε, μια προϊστάμενη αρχή η οποία θα αποφασίζει. Εγώ αυτό θα ήθελα να κάνει η Άζα και θα ήθελα να μάθω εάν ε, προβλέπετε στον κανονισμό σας μια τέτοια δυνατότητα. Ευχαριστώ Τζάκη Φώστα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, καθυστέρησα. Έξι ώρες ε, χρειάστηκε για να έρθω εδώ. Ε, έχουμε απεργία των γεωργών στη χώρα μου. Δύο σημεία θέλω να σχολιάσω. Όταν κάναμε την, τον αρχικό κανονισμό της ΕΑΣΑ, ε, εγώ ήμουν εδώ και για την πιστοποίηση των Α380. Ε, ίσως είμαι μόνη, η μόνη που ήταν τότε εκεί. Είναι αλήθεια ότι τα όσα εμπεριέχει τώρα ο κανονισμός ε, είναι απίστευτα πολλά. Και είναι και η ώρα νομίζω να αντιμετωπίσουμε το πώς θα προχωρήσουμε με το θέμα αυτό. Είμαι πεπισμένη ότι η Άσα έκανε πολύ καλή δουλειά. Ήταν πολύ δύσκολε εποχέ και υπάρχουν λίγα σημεία τα οποία θα ήθελα να σχολιάσω. Θέλω μεγαλύτερη ασφάλεια στον προπολογισμό. Ε, δεν θα μπορούσαμε να περάσουμε σε ένα σύστημα τύπου FAA, αλλά καθώ ο κλάδο ε, δίνει περίπου το 75% των εσόδων ε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση 20 με 25% με 30%, ε, είναι σαφές ότι έχει πολύ ισχυρό ρόλο ο κλάδος να παίζει με πολύ ισχυρό ρόλο στο να διαμορφώσει τον τρόπο λειτουργία τη ΕΑΣΑ. Ε, φυσικά το θέμα των ανεπάνδρωτων αεροσκαφών είναι πολύ σημαντικό και ως συγγήτρια θέλω να δω πώς η συμπερίληψη αυτών των αεροσκαφών θα εξασφαλιστεί στον κανονισμό του ΕΑΣΑ. Θέλω νομίζω να βρούμε μια ε, διεθνή προσέγγιση, να σκεφτούμε φάνταστα, ε, να το κάνουμε καλά ε, σε σχέση με τα σχόλια για το περιβάλλον και την απασχόληση, φυσικά ξέρουμε ποια είναι η εντολή της ΕΑΣΑ και στις της, αλλά η ουσία ποια είναι, ότι θέματα του περιορισμού του χρόνου πτήσης ε, ρυθμίζονται σε επίπεδο εθνικής ε, πολιτικής αεροπορίας ε, και τα παρακολουθούν οι εθνικές αρχές. Και αν υπάρχουν και άλλα θέματα για την απασχόληση, θα ασχοληθούν τα συνδικάτα. Και οι Εθνικέ Αρχέ Πολιτική Αεροπορία θα ασχοληθούν επίση με οποιαδήποτε άλλα θέματα αριθμού πτήσεων, ορών πτήσεων κτλ. Εγώ δεν άκουσα κανένα παράπονο από κανένα από την εισαγωγή τη επικαιροποίηση του FTL. Ούτω ή άλλω, ε, υπάρχει άλλο ένα θέμα που θέλω να θέσω. Διάβασα ένα-δύο πράγματα στο κείμενο σε ό,τι αφορά τον διεθνή ανταγωνισμό, α πούμε και τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Θα πρέπει να συμμορφωθούμε. Περίπου π.χ. για τον ήχο. Θα πρέπει να συμμορφωθούμε με τους κανόνες της ΙΚΑΟ. Δηλαδή να μην θεωρήσουμε ότι μπορούμε να έχουμε ευρωπαϊκούς κανόνες ε, και μετά ε, να μην μπορούμε να συμμορφωθούμε το πράγμα 16, ξέρω εγώ 17 του, της ΙΚΑΟ. Ε, ο ρόλος της ΙΚΑΟ είναι απολύτως σημαντικός και θα πρέπει να απεικονιστεί στο κείμενο όπως πρέπει. Αυτά προς το παρόν από πλευράς μας. Θα συζητήσουμε κάποια από αυτά τα θέματα, είμαι σίγουρη, με περισσότερες λεπτομέρειες. Ευχαριστώ πάντως την Κομισιόν για το σχόλιο της. Α, και ένα τελευταίο που ξέχασα να πω για την ασφάλεια. Γιατί φυσικά από το... Από την 11η Σεπτεμβρίου άλλαξε τελείως το, το, πεδίο. Ε, οι ομάδες ας πούμε, που πηγαίνουν και ελέγχουν ας πούμε, ε, τα αεροπλάνα κτλ. Πώς ασχολούνται με την ασφάλεια. Ε, η Κομισιόν και η ΕΑΣΑ ελπίζουν να βρουν μια κάποια λύση, κάποια, να υπάρξει μια διευθέτηση για το πώς αντιμετωπίζονται αυτά τα θέματα της ασφάλειας στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, συναδέλφοι σας και συνάδελφοι. Θίξαμε πολλά ζητήματα θα ήθελα και εγώ να απευθυνθώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μια ερώτηση γενικού στρατηγικού ενδιαφέροντος σχετικά με το πώς τα μη επανδρομένα αεροσκάφη και η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της ΕΑΣΑ είναι σημαντικά ζητημάτα είναι σαφές, αλλά όταν μιλούμε για μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τον ένα χώρο, η ερώτησή μου θα ήταν κατά πόσον θα είχε νόημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ήταν λίγο πιο φιλόδοξη κατά την προσέγγιση της. Παραδείγματο χάρη, όταν διαβουλευόμαστε για τις φορολογικές βάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή για τους διαφορετικούς χρόνους δραστηριότητας, επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ευρώπη. Επειδή τη σύγκριση θα διαπιστώσουμε μια πολύ πιο περιοριστική πολιτική στην Ευρώπη. Αλλά ως σοσιαλδημοκράτη θα ήθελα το θέμα αυτό να προσεγγιστεί για άλλη μια φορά από ευρωπαϊκή προοπτική. Και αυτό που μου λείπει επίσης στη δεσμή μέτρων είναι πως δεν έχουμε μια πολιτική υποδομών της ευρωπαϊκής αεροπορίας όπως θα την έλεγα. Όλα γίνονται σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο αλλά όχι σε ευρωπαϊκό. Δεν γνωρίζουμε λοιπόν σε ποια σε ποια κατεύθυνση θα κινηθούμε τα επόμενα δέκα έτη ως προς τις υποδομές ή που θέλουμε να γλύξουμε. Αυτή θα ήταν πρώτη μου ερώτηση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φοβήθηκε ίσως, δίστασε να ληξουμε αυτη θα ηταν η πρωτη μου ερωτηση γιατι η ευρωπαικη επιτροπη φοβηθηκε ισως διστασε να ακουμπησει την καυτή πέτρα της αρμοδιότητας των εθνικών αρμοδιοτήτων και μια και μιλάω για εθνικές αρμοδιότητες επιτρέψτε μια δεύτερη ερώτηση αφότου μιλήσουμε για την διεύρυνση αρμοδιοτήτων της ΕΑΣΑ θα με ενδιαφέρε πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να χωρίσει περαιτέρω αρμοδιότητες στην ΕΑΣΑ όσον αφορά την ασφάλεια και το περιβάλλον. Αυτό γίνεται σε διαφορετικά επίπεδα. Θα με ενδιαφέρε κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να φανταστεί να διευρύνει τις αρμοδιότητες της ΕΑΣΑ προς αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πάρα πολύ μια παρατήρηση για τις εθνικές αρμοδιότητες. Στη Γερμανία θα χαιρόμασταν εάν υπήρχε μια εθνική αρμοδιότητα για τον εναέριο χώρο. Εκεί έχουμε 16 αρμοδιότητες των ομόσπονδων κρατηδίων τα οποία αποφασίζουν για την ανοικοδόμηση ενός αεροδρομίου. Αν μιλούμε για το ευρωπαϊκό επίπεδο είναι μια πολύ καλή ιδέα αλλά και στις χώρες μας θα πρέπει να εργαστούμε για να υπάρχει μια εθνική αρμοδιότητα όπως υπάρχει στην οδική κυκλοφορία. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει στην αεροπορία και στην αυσιπλοεία. Και στα τα εξωτερικά σύνορα είναι συναρμόδια 5-6 υπουργεία επιπρόσθετα στα ομόσπονδα κρατήδια αλλά φυσικά και θα ήταν σωστό να πάμε προς την ευρωπαϊκή κατεύθυνση. Έχουμε ένα σωρό ερωτήσεις. Φυσικά και χαρήκαμε για την πρότασή σας. Τώρα έχετε τη δυνατότητα να εκφραστείτε κύριε Κορνέλιος, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όντως έχουν ανακύψει πάρα πολλά θέματα. Χαιρόμαστε βέβαια για το ενδιαφέρον, για την πρόταση αυτή, το οποίο υπόσχεται πολλά για τις επερχόμενες συζητήσεις μαζί σας και τις οποίες χαιρόμαστε. Η πρώτη ομιλήτρια, η κυρία Μαρινέσκου, χαιρόμαστε πολύ, σας συγχαίρουμε που θα είστε η εισηγήτρια όσον αφορά τα ζητήματα που, ανεφ, που αναφέρθηκαν, πρώτα απ' όλα το όνομα της ΕΑΖΑ. Πιστεύω πως ένα από τα καλύτερα επιχειρήματα για τη διατήρηση του ονόματος είναι πως, πρόκει, πως είναι αρκετά γνωστό σε όλο τον κόσμο και κανονικά όταν έχει κανείς ένα όνομα σαν μια, ένα εμπορικό σήμα αυτό λειτουργεί. Γι' αυτό και δεν βλέπουμε κανέναν λόγο να αποποιηθούμε το όνομα αυτό. Αναφερθήκατε στα μη επανδρομένα αεροσκάφη, πολλοί άλλοι επίσης αναφερθήκαν στα αεροσκάφη αυτά, θα επανέλθω στο θέμα αυτό. Όσον αφορά τα πρόστιμα και τις κυρώσεις, υπάρχουν κάποια ποσοστά στον κανονισμό, θα, θα βρούμε εκεί τα μέγιστα πρόστιμα και τις μέγιστες κυρώσεις. Δεν αλλάξαμε κάτι, υπάρχουν στον επικαιρό κανονισμό και είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως πρόκειται για το τελευταίο μέτρο, δηλαδή δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ μέχρι στιγμής. Υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι για να διασφαλίσουμε μια καλή συμμόρφωση με τους κανόνες και κάποιες φορές το να χρησιμοποιούμε αποτρεπτικά ένα αυστηρό μέτρο βοηθάει στην συμμόρφωση με τους κανονισμούς. Η διεθνή συνεργασία αναφέρθηκε από τον κύριο Μαρουνέσκο μεταξύ ΕΑΖΑ και πολιτιών Έχουμε κάποια πρόοδο εκεί. Είχαμε κάποιες ζημερείς συναντήσεις πριν από δύο εβδομάδες με τις ΗΠΑ και επιτύχαμε για πρώτη φορά μια συμφωνία σύμφωνα με την οποία κάποια μικρά προϊόντα δεν θα χρειάζονται πλέον πιστοποίηση. Σε καμία από τις δύο κατευθύνσεις, για κάποια άλλα προϊόντα συμφωνήθηκε πως θα υπάρχει μια απλή διοικητική διαδικασία, ένα απλό έγγραφο που θα πρέπει να έχει υπογραφεί και έτσι θα μειώσουμε τα έξοδα για τη βιομηχανία και συμφωνήσαμε επίσης με τις ΗΠΑ να προσπαθήσουμε να μειώσουμε την διπλή εργασία από τις δύο πλευρές όσον αφορά την πιστοποίηση των μεγάλων αεροσκαφών των δύο πλευρών. Όσον αφορά την ασφάλεια security, η κυρία Πρόεδρε και ο κ. Μαρινέσκου αναφέρθηκαν στο ότι φυσικά και χρειαζόμαστε την ικανότητα να ασχοληθούμε με ζητήματα ασφάλειας, τέθηκε το ζήτημα ποιος είναι ο ρόλος της Επιτροπής ως προς την ΕΑΣΑ και σε σχέση με τα κράτη-μέλη. Εμείς διασανόμαστε πως ο καθένας έχει τον ρόλο του και το κείμενο που προτείναμε εδώ περιέχει κάποια στοιχεία παραπάνω, ειδικότερα στην δύναμη συμβολή της ΕΑΣΑ σε ζητήματα ασφάλειας παραμένοντας ωστόσο ο καθένα στον τομέα τη τεχνογνωσία του. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι στον τομέα του σχεδιασμού αεροσκαφών η πραγματική τεχνογνωσία υπάρχει από την πλευρά της ΕΑΣΑ όσον αφορά την ασφάλεια, παραδείγματος χάρη την κυβερνοασφάλεια από πολλές απόψεις. Η ΕΑΣΑ πρέπει να αποτελεί μέρος των λύσεων. Αλλά επίσης υπάρχουν περιπτώσεις παραδείγματο χάρη ω προ την πρόσβαση σε πληροφορίε, η οποία είναι καθοριστική σημαντική και έχουμε υπηρεσίες ασφάλειας, πληροφοριών. Πρέπει να συνεργαζόμαστε λοιπόν και το κάνουμε με ευχαρίστηση. Συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να επιτύχουμε όσο δυνατόν περισσότερες κοινέ αξιολογήσεις κινδύνου και να λάβουμε μέτρα είτε με ένα νομικό θεμέλιο ασφάλειας ή υπό ένα εθνικό νομικό θεμέλιο. Στην τομέα των περιοχών συγκρούσεων που αναφέρθηκε από κάποιους προσπαθούμε να κάνουμε ακριβώς αυτό. Να αλληλοσυμπληρώνονται όλοι όσοι μπορούν να συμβάλλουν και συγκεκριμένα να προσπαθήσουμε να πετύχουμε την καλύτερη κοινή αξιολόγηση μέσω συνεργασία των κρατών μελών. Έχουμε τη γνώση και στη συνέχεια πρέπει να βρούμε τον τρόπο να επικοινωνήσουμε την, τις πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο σε όλους τους αερομετοφορείς επειδή πιστεύουμε πως πληροφορίες σημαντικές για την ασφάλεια πρέπει να διατίθενται και δεν θα πρέπει να περιορίζονται σε έναν ή δύο αερομεταφορείς καθώς οι Ευρωπαίοι πολίτες ταξιδεύουν με όλες τις αερογραμμές και όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να προχωρήσω με τα ζητήματα της που έθεσε η κυρία Πρόης, ανέφερε όπως και πολλοί άλλοι το ζήτημα του προϋπολογισμού της ΕΑΣΑ, την ανάγκη να παραμείνει να παραμείνουν διαθέσιμοι οι οικονομικοί πόροι, η διατήρηση της ευελιξίας. Πιστεύω πως το λάβαμε υπόψη το ζήτημα αυτό στην πρόταση. Εσείς θα το κρίνετε. Εμείς ωστόσο αναμένουμε με χαρά την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με αυτό προσθέσαμε τη δυνατότητα ή μάλλον κάποια στοιχεία όπως τους δείκτες που ανέφερα, δείκτες φόρτου εργασίας που θα σας βοηθήσουν εσάς και το Συμβούλιο κατά την εκπόνηση του προ... ετήσιου προϋπολογισμού για το σωστό επίπεδο προσωπικού για την υπηρεσία έτσι ώστε αυτή να μπορεί να κινείται στην αγορά και να μην καθυστερεί κατά την πιστοποίηση με τη ε, καθυστέρηση πρέπει να αποφεύγεται για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας. Επίσης αναφέρθηκε ο ενεργός διεθνής ρόλος που μπορεί να παίξει η ΆΣΑ. Χρειαζόμαστε τους πόρους, την νομική βάση και πιστεύουμε πως αυτή η πρόταση εμπεριέχει και τα δύο. Έτσι ώστε η ΕΑΣΑ θα μπορέσει να μας βοηθήσει να εξάγουμε ευρωπαϊκά πρότυπα ώστε να βοηθήσουμε χώρες του τρίτου κόσμου να βελτιώσουν την ασφάλεια Τίποτα δεν εμποδίζει την παρουσία της ΕΑΣΑ σε τρίτες χώρες, ήδη είναι παρουσία εκεί. Παραδείγματο χάρη η ΕΑΣΑ μας βοηθάει τώρα πολύ με τεχνικές εργασίες. Αποκινούμε την Κίνα για να τεθούν τα θεμέλια για, ένα, για μια μελλοντική συμφωνία ασφάλειας αεροπορίας αυτή η δραστηριότητα της ΕΑΣΑ σε διεθνές επίπεδο είναι αναγκαία, σαφώς, και προωθείται σε διεθνή φόρουμ. Η ΕΑΣΑ είναι επίσης παρούσα. Είναι παρούσα ως μέρος της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως, ως παρατηρητής στα περισσότερα σώματα της ΕΚΕΟ, Επίσης σε τεχνικές ομάδες, παραδείγματο χάρη, προεδρεύει ένα πάνελ της ΕΙΚΕΟ, αυτό που ασχολείται με αεροσκάφη συγκεκριμένα. Ο κύριος Βαντάλεν αναφέρθηκε στον ρόλο της ΕΑΣΑ σε σχέση με τις εθνικές αρχές και ποιος διατηρεί την τεχνογνωσία για τις επιθεωρήσεις. Αυτό εξαρτάται από τους διαφορετικούς κανόνες που έχουν οι ΕΑΣΑ και οι εθνικές αρχές. Σε κάποιες περιπτώσεις η ΕΑΣΑ δικαιούται να είναι αρμόδια, όπως παραδείγματος χάρη στον τομέα της πιστοποίησης αεροσκοφών, αλλά σε άλλους τομείς αυτό δεν ισχύει καθόλου. Παραδείγματος χάρη, όσον αφορά τους κανόνες επιχειρησιακής ασφάλειας, εκεί η αρμοδιότητα βρίσκεται στις εθνικές αρχές, οι οποίες στέλνουν τους επιθεωρητές, τους κατάλληλα καταρτισμένους επιθεωρητές, επίσης μπορούν να χειρώσουν τέλη για αυτό. Αυτό που προτείναμε εμείς ως προς αυτό, έτσι ώστε τα μέτρα αυτά να αποκτήσουν ένα πιο ενιαίο πρόσωπο, είναι κάποιες βασικές προϋποθέσεις για τους επιθεωρητές ασφάλειας και τη δυνατότητα μιας στενότερης συνεργασίας των κρατών μελών, έτσι ώστε να γίνεται σε κάποιες φορές μια ανταλλαγή υψηλώς καταρτισμένων επιθεωρητών. Ο κ. Βαν Μίτεμποχ ενημερώθηκε για τη δυνατότητα κατάρτισης πιλότων μη επανδρομένων αεροσκαφών. Η πρόταση την οποία εκπονήσαμε δεν είναι τόσο αναλυτική. Αυτό πιστεύω πως θα πρέπει να εξαρτάται από το, την επικινδυνότητα της επιχείρησης. Μέτρα θα ληφθούν αργότερα στα οποία θα αποφασιστεί σε ποια περίπτωση θα πρέπει να απαιτείται κατάρτιση και σε ποια όχι. όσον αφορά την αλλαγή και την καινοτομία που τέθηκε από την κυρία Κίνονεν. Πιστεύω πως βελτιώσαμε τις δυνατότητες. Πιστεύω ότι αυτή η πρόταση έχει λιγότερες προδιαγραφές, είναι πιο ευέλικτη και πιστεύω πως θα μας βοηθήσει τα επόμενα 10-15 χρόνια να έχουμε ένα επαρκές νομικό θεμέλιο. Η κυρία Ντέλη αναφέρθηκε στο ερώτημα της αύξησης των εκπομπών αυτό δεν αποτελεί θέμα μόνο αυτής της πρότασης, σε κάποιο βαθμό βέβαια ναι. Εδώ δουλεύουμε με, μια, με την προσέγγιση μια δέσμης μέτρων, τα οποία μέτρα θα πρέπει να μας βοηθήσουν να κρατήσουμε τις εκπομπές χαμηλές. Ένα από, μία από τις πτυχές είναι οι τεχνολογίες, και εκεί μπαίνει στο παιχνίδι η Άσα, η οποία θα μας βοηθήσει να εφαρμόσουμε Τις τεχνικές λύσεις. Υπάρχουν ωστόσο και άλλα ζητήματα, όπως επιχειρησιακά μέτρα αεροπορίας, τα καύσιμα και φυσικά μηχανισμοί της αγοράς για να καλύψουμε το κενό. Και όπως γνωρίζετε εργαζόμαστε πολύ σκληρά για να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε στην συνέλευση της ΕΚΕΟ μια παγκόσμια συμφωνία για, μια, για έναν κοινό παγκόσμιο μηχανισμό της αγοράς αντικρώμενα συμφέροντα. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί που αφορούν την ΕΑΖΑ και το Διοικητικό Συμβούλιο, που είναι πολύ συγκεκριμένοι. Για την υγεία των πιλότων, πολλοί αναφέρθηκαν στην πτήση της German Wings. Η ΕΑΖΑ έχει αναπτύξει πολλές συστάσεις μετά από αυτό το συμβάν και Προετοιμάζεται τώρα η εφαρμογή τους και οπωσδήποτε θα το προωθήσουμε το θέμα μαζί με την ΕΑΖΑ ήδη φέτος. Στην πρόταση αυτή συγκεκριμένα έχουμε αυξήσει ιδιαίτερα τις πιθανότητες ανταλλαγής δεδομένων και ιατρικών δεδομένων. Είναι όμως πολύ δύσκολο το θέμα, αλλά θεωρούμε πως έχουμε μια σωστή νομική βάση. Η κυρία Γιάλα Σέντερ νομίζω ανέφερε την έδρα της ΕΑΖΑ ναι, αναφέρουμε ότι η κολονία είναι στον κανονισμό και η ΑΖΑ νομίζω μαζί με τη Γερμανία έχουν προχωρήσει όσον αφορά τη συμφωνία εγκατάστασης. Ο ανθρώπινος παράγων είναι πάρα πολύ σημαντικός και προβλέπεται ε, η υπομορφή εκπαίδευση των πιλότων, ιατρικών πιστοποιητικών, αλλά πρέπει να τονίσω ότι και άλλοι τομείς, όπως περιορισμοί χρόνου ζητήματα συμβάσεων. Όπως μάθαμε από την ε, έκθεση για το συμβάν της German Wings δεν είχαν άμεση σχέση. Ο κύριος Φάντεκάμπ ανέφερε τον προπολογισμό. Το κάλυψα ήδη νομίζω. Προσπαθώ να είμαι σύντομος, όπως μου είπατε κύριε Πρόεδρε. Μη επανδρομένα αεροσκάφη και ασφάλεια Τώρα, εάν η ΑΖΑ θα πρέπει να έχει μια πιο έντονη εντολή, νομίζω το κάναμε αυτό. Υπάρχει μια ολοκληρωμένη αγορά με αμοιβαία αναγνώριση και αυτό απαιτεί και αμοιβαία υποπτία. Και μια καινοτομία αυτής της πρότασης είναι ακριβώς ότι η ΑΖΑ πέρα από τα καθήκοντα που ήδη έχει μπορεί να αναλάβει τα καθήκοντα εάν το επιθυμούν ε, τα κράτη-μέλη. Ε, αν ενδιαφέρονται να έχουν, αν δεν ενδιαφέρονται να έχουν επιθεωρητές για τη χύψη δραστηριότητα, μπορούν να το αναθέσουν στην ΕΑΖΑ, κάτι το οποίο σήμερα δεν είναι δυνατόν. Η κυρία Φώστερ βεβαίως αναφέρθηκε στην έκθεσή της για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, ε, για την οποία την ευχαριστούμε και νομίζω πως θα συμφωνήσει πως η πρότασή μας συμφωνεί με τα συμπεράσματα της έκθεσής της. Και τέλος ο κύριος Ερτούγ ε, αναφέρθηκε στον πως θα πρέπει να είμαστε κάπως πιο φιλόδοξοι. Ανέφερε ζητήματα όπως οι διαφορές στην φορολογία, κανόνες χρονοεργασίας ε, σε τρίτες χώρες. Είναι ζητήματα που υπάρχουν ε, στην στρατηγική της αεροπορίας, αλλά ίσως δεν αφορούν το πεδίο εφαρμογή αυτού του κανονισμού εδώ πέρα. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε όσον αφορά την εξαγωγή ευρωπαϊκών προδιαγραφών είναι ακριβώς να είμαστε δραστήριοι στον ΙΚΑΟ και μέσω διμερών συμφωνιών ε, για την αεροπορική ασφάλεια όπως έχουμε με ΙΠΑ, Βραζιλία, Καναδά και για τις οποίες λάβαμε πρόσφατα εντολή για να διαπραγματευτούμε κι άλλες με την Κίνα και την Ιαπωνία. Αυτά ήταν τα βασικά. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ναι, κύριε Πρόεδρε, θέλω μια συγκεκριμένη απάντηση που δεν έλαβα για το ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η άποψη του προσωπικού, πιλότων και μη, για ζητήματα απόδοσης και κινδύνου. Και ποια είναι η δικαιολογία, η αιτιολόγηση για το ότι φεύγουμε από πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές που είχαμε. Σύντομα παρακαλώ. Είναι σημαντικό γιατί μίλησα βεβαίω για κανόνες που βασίζονται στα αποτελέσματα. Αυτό είναι το νέο στοιχείο. Δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε πολύ συγκεκριμένους ε, κανόνες που θα καθορίζουν ε, τα πράγματα. Είναι πολύ συγκεκριμένοι αυτοί οι κανόνες όσον αφορά π.χ. τον περιορισμό χρόνου πτήσης και υπάρχουν λόγοι να μείνουν έτσι. Ε, αυτό το οποίο προτείνουμε λοιπόν εδώ πέρα είναι να βασιζόμαστε περισσότερο σε κανόνες ε, με βάση την απόδοση, όπου αυτό είναι η καλύτερη μέθοδος, χωρίς αυτό να σημαίνει πως είναι πάντα η καλύτερη μέθοδος. Μάλιστα, ευχαριστώ, τελειώσαμε, περνάμε στο επόμενο σημείο πρωτόκολλο τροποποίησης ε, της ε, Συμφωνίας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ισραήλ και την Κροατία για να ληφθεί υπόψη η ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε τον λόγο, κύριε Ε, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα δύο ταυτόσιμα νομοθετήματα. Το ένα αφορά την ένταξη της Κροατίας και έχουμε συστάσεις από το Συμβούλιο σύμφωνα με την κοινή πολιτική, την κοινή συμφωνία με την Γεωργία και η ίδια ακριβώς ε, περίπτωση πρόκειται για την Ευρωμεσογειακή Αεροπορική Συμφωνία με το Ισραήλ. Δεν υπάρχουν λάγες στην συμφωνία, στις συμφωνίες και τις δύο, και με τη Γεωργία και με το Ισραήλ. Καμία ουσιαστική αλλαγή. Η μόνη αλλαγή είναι η συμπερίληψη της Κροατίας λόγω της ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ντελή, ευχαριστώ. Είναι τεχνικά αυτά τα θέματα. Όσον αφορά την επέκτασή τους δηλαδή για να καλύπτουν και την Κροατία συμφωνίες που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ και τη Γεωργία. Οπότε δεν θα πω τίποτα άλλο. Είναι τεχνικά ζητήματα. Πρέπει να υπερψηφίσουμε νομίζω στην Ολομέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τζάκι Φώστερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Προφανώς <laughs> δεν είναι δύσκολα πράγματα. Ας τελειώνουμε με αυτές τις συμφωνίες. Υπάρχουν και άλλες συμφωνίες που περιμένουν. Οπωσδήποτε το ECR θέλουμε να προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Ευχαριστώ, Ράντος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. εξ ονόματος της Άλντε υποστηρίζουμε την συμφωνία όσον αφορά την ένταξη της Κροατίας. Η Κροατία έχει υπογράψει το 98 συμφωνία αεροπορική με το Ισραήλ στο πλαίσιο τουριστικών συμφωνιών. Τώρα εδώ πέρα έχουμε απλοποιημένη διαδικασία για καλύτερη οικονομική συνεργασία με το Ισραήλ, ειδικά στον τομέα του τουρισμού. Αυτά σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Προθεσμία είναι, για τις τροπολογίες είναι 21 Μαρτίου στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Παρακαλώ να τηρηθεί. Και περνάμε στο επόμενο θέμα. Η συμφωνία με την Γεωργία. Και πάλι έχουμε τροποποιήσει λόγω της ένταξης της Κροατίας. Και πάλι εδώ πέρα ο εισηγητής έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόκειται για το ίδιο ακριβώς πράγμα σε αυτό το κείμενο. Μιλήσαμε μόλις τώρα για μια συμφωνία με το Ισραήλ. Τώρα εδώ έχουμε μια συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της και της Γεωργίας. Ίδια απόφαση είναι αυτή. Αλλάζει η χώρα. Είναι μια απόφαση που πρέπει να υιοθετήσουμε μετά από την προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ. Ντελή, εκ μέρους του ΕΡΚ, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε την Κροατία το συντομότερο δυνατόν και σε αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστώ. Ε, συμφωνώ. Υποστηρίζουν οι συγητή, λέει η κυρία Φώστερ. Ο κύριος Ευχαριστώ. Εμείς δεν είχαμε συμφωνία συνεργασίας στην Κροατία, δηλαδή εμείς στην Κροατία με την ε, Γεωργία, άρα θα πρέπει να περάσει αυτή η συμφωνία. Υιοθετείτε. Κλείνει. Η μοναδική δυνατότητα τροποποίηση είναι η απόρριψη. Αλλά άλλε αιτήσει δεν θα ήταν παραδεκτέ. Ωραία. Αυτό θα ήταν το τέλος του δημόσιου μέρους της συνεδρίασης. Περνάμε στη συνεδρίαση και κλεισμένο των θυρών. Αλλά τώρα θα ήθελα να παρακαλέσω αυτούς που δεν τους επιτρέπεται να βρίσκονται εδώ να εγκαταλείψουν την έσοδα, την αίθουσα. Όλοι οι βουλευτές μπορούν να παραμείνουν.